Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούχνερ εκ μέρους των Πρασίνων. Όχι, δεν έχετε σχόλιο. Κυρία Μπαγκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε, κάπως με ξέπηξε το ότι δεν μίλησε κανείς σήμερα για την γνωμοδότηση του συνάδελφου Όμπερμαγερ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική από πλευράς περιεχομένου θέλω να πιστεύω, δεν υπάρχει κάποιο είδους προκατάληψη όσον αφορά τη δουλειά μιας κοινοβουλευτική ομάδας εκεί όπου ανοίγει και η ε, κυρία Λεπέν. Και εμείς συμμετέχουμε ε, σε αυτή την πολιτική ομάδα. Ε, αλλά πάντως πάνω απ' όλα είναι το δικαίωμα των πολιτών, το δικαίωμα τους να ακούγονται στα πλαίσια των ε, θεσμικών οργάνων και ελπίζω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση σαμποταρίσματος του συναδελφού ε, είτε ως προσωπική αιχμή είτε ως πολιτική ομάδα γιατί κάποιοι πολίτες ψήφισαν αυτή την πολιτική ομάδα αυτό θα ήταν πάρα πολύ αντιπαραγωγικό το μόνο το οποίο θα γινόταν θα ήταν θα αυξανόταν δυσφορία κατά κατά της Ευρώπης. Μα αυτό είναι σαν της δικτατορίας. Εκεί ε, δεν υπάρχει ευθεία του λόγου και δεν συμφωνούμε με αυτό. Η έκθεση είναι πάρα πολύ ισορροπημένη. Τονίζεται η σημασία της συμμετοχής των εθνικών ε, ε, κοινοβουλίων και όσον αφορά τις ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και νομίζω ότι όντας τόσο αξιόλογη αυτή η έκθεση θα αξίζει να συζητηθεί. Ο πρόεδρος ευχαριστούμε εμείς και δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για τη δουλειά που έκανε κατά την προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά την ε, δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο και την προθυμία που έχει δείξει να ασχοληθεί με το θέμα. Η Επιτροπή σας έχει συνεργαστεί πολύ καλά και έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή και με εμάς αλλά και εμείς με τα Εθνικά Κοινοβούλια και προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς αυτά μπορούν να συνεισφέρουν. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και είναι όπως ε, αναφέρεται και στο σχέδιο έκθεσης εξίσου σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες. Τα κοινοβούλια λοιπόν έχουν επαρκή πληροφόρηση μέσω των κυβερνήσεων, μέσω των εκπροσώπων του στο Συμβούλιο και οι πληροφορίες αυτές ε, να τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν τον θεσμικό τους ρόλο. Και σε θέματα πολιτικής επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξει το ρόλο και υπάρχουν ορισμένα θέματα στα οποία υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Η έκθεση αυτή θα επικεντρωθεί στο εμπόριο και φυσικά θα καλωσορίσουμε την ε, συνεισφορά σας. Είμαστε έτοιμοι για συζήτηση και θέλουμε να αυξηθούν οι προσπάθειες για την ε, δυσφάλιση της διαφάνειας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Ομπερμάιρ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Ο συνάδελφος κύριος Καρίμ μας έφερε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα και νομίζω πως τα επιχειρήματά του ήταν αρκετά καλά και Σίγουρα δεν ε, αποκάλυψε όλες τις πληροφορίες, όμως είμαι σίγουρος ότι και αυτό σκέφτεται τις εκλογές, σκέφτεται τους ψηφοφόρους του, ξέρει τι κάνει. Εγώ είμαι αισιόδοξο. έχω νομίζω μια καλή πρόθεση, είμαι αισιόδοξο ότι θα υπάρξει πρόοδος. και ελπίζω να υπερβούμε τα πολιτικά και τα κομματικά ε, συμφέροντα και να οδηγηθούμε σε μια λύση η οποία θα γίνει αποδεκτή από τα κράτη-μέλη, θα γίνει αποδεκτή από τους πολίτες και θα γίνει όχι μόνο αποδεκτή αλλά και καλύτερα ανεκτή. Είναι σίγουρα προς το συμφέρον όλων να υπερβούμε τις ε, πολιτικές μας ε, διαφορές. Τώρα το κείμενο είναι σε γενικές ε, γραμμές εντάξει, ωστόσο θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία, να κάνω κάποια σχόλια. Μας λέτε ότι πρέπει να ε, συμμετέχουν πιο ενεργά οι κυβερνήσεις των ε, κρατών μελών. Πώς όμως ακριβώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάποια δομή κάποια διαρθρω... κάποιος ε, διαρθρωμένος ε, διάλογος. Επίσης αναφέρεστε στην συνεργασία με τις μη κυβερνικές οργανώσεις και εδώ θα ήθελα να ακούσω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Α, ναι, λοιπόν, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ... τοπολογιών στις 21 Ιουνίου, 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 24. Μία ανταλλαγή απόψεων για την συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Εξυγχρονισμός της ε, συμφωνίας αυτής. Εδώ Έχουμε δύο σχέδια έγκρισης, δύο σχέδια έκθεσης να εγκρίνουμε. Σήμερα συναντήσαμε τον κύριο Ραούλ Φερνάντες και τον καλέσαμε. Είναι εδώ στην Επιτροπή, πρέσβης της Δημοκρατίας της Χιλής και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ροντρίγκε Πινέρο. Λείπει όμως. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να την αντικαταστήσει και να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσω τότε το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, τον κύριο Μάτο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η η Μακουλάδα Ροντρίγκε Πινιέρο απουσιάζει δυστυχώ, όμω έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ το θέμα αυτό. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον πρέσβη. Συμφωνούμε απόλυτα με το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστή η βιολογική παραγωγή, να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων αυτών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Είχαμε θέματα συντονισμού, ακριβώς γιατί τρέχουν δύο παράλληλες εκθέσεις. Πρώτα η εκθέση για τον πυλώνα του εμπορίου. Εδώ διεξάγονται τριμερείς διάλογοι για τον κανονισμό για τα βιολογικά προϊόντα, τη βιολογική γεωργία και ανάλογα το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου θα γίνουν πολλές τροποποιήσεις, πολλές αλλαγές στη Γενική Συμφωνία. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω πως ε, θα επηρεάσει και τον κανονισμό. Εδώ πρέπει να νομοθετήσουμε σύμφωνα με τις ε, προδιαγραφές. Και το παρακολουθούμε γιατί υπάρχει φόβος ο πλευρά των Ευρωπαίων ε, Γεωργών. Δηλαδή, μιλούμε τώρα για ισοδυναμία και φαίνεται κάπως αντιφατικό ότι σε κάποιες χώρες ή το σε κάποιες περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποιες ουσίες για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, αλλά να μην επιτρέπεται αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχει εδώ δυσμενής διάκριση και θα πρέπει αυτό να αποφεύγεται. Επίσης, να ληφθεί υπόψη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκθεση της ε, υπηρεσίας για την ε, για τα είδη διατροφής και την υγεία και από κάποιους άλλους ε, φορείς πιστοποίησης για να δούμε το τι θα ισχύει με τις εξαγωγές. Θεωρούμε θετική αυτή τη συμφωνία, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι σημαντικός ε, εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωση η Χιλή. Οπότε θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε αυτή τη ε, συμφωνία. Και να δούμε τι θα γίνει με κάποιες τροπολογίες που μας ε, ανησυχούν. Όχι από πλευράς ουσίας, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα όπως με τις κυρώσεις. Δεν θα πρέπει να ισχύσει σύστημα κυρώσεων όπως αναφέρεται στην αιτιολογική παραγραφό G. Θεωρούμε ότι δεν είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε παραδείγματα όπως με τις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδείχθηκε ότι δεν αποδίδουν, δεν ωφελούν αυτές οι κυρώσεις. Καλύτερα συνεργασία και διάλογος παρά κυρώσεις. Και κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί είναι το άρθρο λάμδα που αφορά τους αποσπασμένους εργαζομένους. Θα πρέπει εδώ να γίνει μια διάκριση για το ποιους εργαζομένους καλύπτουμε εδώ. Μήπως και εδώ είναι υπερβολικό να θέλουμε να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία εν προκειμένου. Πάντως συμφωνούμε με την τροπολογία π και θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε κάποιες υποχρεώσεις που ισχύουν για όλες τις χώρες. Δηλαδή για τις αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών. Συνεχίζονται οι διοραματεύσεις για το θέμα. Άρα δεν είναι σωστό να επιβάλλουμε στην Χιλή μια τέτοια υποχρέωση, αφού αυτή η υποχρέωση δεν έχει υιοθετηθεί για εμάς τους ίδιους ακόμα εδώ στην Ευρώπη. Καταβάλει σοβαρές προσπάθειες η Χιλή για να προχωρήσει το θέμα της ισότητα των φύλων. Α, δεν ξέρω τώρα αν χρειάζεται να υπάρχει στην ε, ε, συμφωνία, αν χρειάζεται ιδιαίτερο κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατοχυρώσουν την ισότητα των φίλων. Ίσως δεν χρειάζεται το ξεχωριστό κεφάλαιο. Για κάποια άλλα δευτερεύοντα θέματα θα τα πούμε. Πάντως πάρα πολύ θετική αυτή η πρόταση αναγκαία και έτσι με κάποια αδελφή χώρα θα αναβαθμίσουμε θέσεις της χώρας και για μας βέβαια ακόμα καλύτερα που είμαστε Ισπανία. Άρα χωρίς επιφυλάξεις θα εγκρίνουμε την πρόταση. Ευχαριστώ λίγο πρόεδρος, θα δώσω τώρα το λόγο στον πρέσβη. Κύριε Φερνάντες. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντιμος. Ευχαριστώ που με καλέσατε για να συζητήσουμε και συμφωνώ με τόσο που ο κύριος και υπάρχει ένα σημαντικό σημείο πάντως για μας πρώτα-πρώτα όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Έχουμε καταβάλει σημαντική προσπάθεια ούτω ώστε να φτάσουμε σε κάποια πρότυπα και έτσι να μπορούμε να έχουμε αμοιβαιότητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής θα υπάρξει αμοιβιότητες. Αυτό είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Και γι' αυτό και εμείς τιμούμε αυτήν την συμφωνία. Θα γίνει η προσπάθεια εναρμόνισης, ξεκίνησε από το 2002 που είχαμε την προηγούμενη ε, συμφωνία με την Ένωση σήμερα. επομένω θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε, να προσαρμόσουμε κάποια κομμάτια της συμφωνίας, κάποια κομμάτια τα οποία ήταν στην τότε. Αλλά σήμερα μιλούμε για την κυκλική οικονομία, μιλούμε για ένα σημαντικό στοιχείο όπως η βιώσιμη ανάπτυξη. Μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να καλυφθούν. Και χαίρομαι πολύ ξεκίνησε αυτή η διαπραγμάτευση. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Και τώρα. Έχει το λόγο η συγκεντρία μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. συμπαθάτε με είχα μια άλλη υποχρέωση στις 4.30 και τέλος πάντων θερμούς χαιρετισμού που να στείλω στην πρεσβεία της Χιλής, τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε την ε, στενή μας συνεργασία για να εξασφαλίσουμε τις καλές εμπορικές σχέσεις με την χώρα αυτή. Δεν μπόρεσα να ακούσω ε, την άποψη του συναδέλφου από την Επιτροπή Γεωργίας. Πάντως ε, στην Επιτροπή Γεωργία είχαμε πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία για την έγκριση του κειμένου. Τώρα όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Ε, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, το δώσαμε προτεραιότητα γιατί θεωρούμε ότι ε, τηρούνται όλα τα πρότυπα, υπάρχουν όλε οι εγγύσει ελέγχου για την βιολογική παραγωγή και υπάρχει η αμοιβαιότητα στην πιστοποίηση. Αναγνωρίζει όλα τα πιστοποιημένα μας προϊόντα η Χιλή. Εμείς ε, εξαιρούμε κάποια ζωικά ε, προϊόντα και επίσης κάποια προϊόντα χθιοκαλλιέργειας. Επίσης ε, είναι σημαντικό ότι κανένα χιλιανό προϊόν μπορεί να θεωρηθεί βιολογικό εάν έχει μέσα κάποιες ουσίες από τρίτες χώρες που δεν τις αναγνωρίζουμε όσον αφορά την ισοτιμία. Και επίσης, αν οι έλεγχοι το δείξουν, επίσης υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και εποπτεία για αυτή τη συμφωνία και βέβαια αν χρειαστεί θα αλλάξει ο κατάλογος των προϊόντων. Και οπότε, λαμβάνοντα υπόψη τη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής Γεωργίας, ε, προτείνω να εγκρίνουμε την ε, συμφωνία. Κατά τι διαπραγματεύσει υπήρχε έλλειμμα πληροφόρηση, οπότε παρακαλώ η Επιτροπή να ενημερώνει και το Κοινοβούλιο και τους άλλους ενδιαφέροντες και επίσης να μας ενημερώνει για, την, για, ε, ε, για τις εργασίες της κοινή Επιτροπής. Είπαμε ότι θέλουμε να δούμε κατά πόσο είναι σωστή η παρέκταση αυτής και επέκταση αυτής της συμφωνίας και με ότι κάθε τρία χρόνια γίνεται σχετική αξιολόγηση. Ε, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας που φτάσαμε σε αυτή τη φάση να προτείνουμε την ε, έγκριση της συμφωνίας. Τώρα έχουμε συγχρονισμό του τρίτου πυλώνα συμφωνία σύνδεση ΕΕ Χιλή. Έχουμε εδώ πέρα ένα χρονοδιάγραμμα που είναι πάρα πολύ πιεστικό, πάρα πολύ στενό, γιατί έχουμε τη κοινή επιτροπή, ε, τι προτάσει. Οπότε θα πρέπει να προτείνουμε τι δικέ μα ε, θέσει πριν εγκρίνει τι καθημερινέ γραμμέ ε, το Συμβούλιο. Είναι, είναι εταίρος ε, ιδιαίτερα σημαντικός στα πλαίσια ε, των προστασίας των οποίων δικαιωμάτων και για τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση. Οπότε αυτή η συμφωνία του 2002 έχει λειτουργήσει καλά, έχουν διπλασιαστεί οι εμπορικέ ροέ, ε, έχουν αυξηθεί οι επενδύσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγει ωφελημένη. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό αυτής της ε, συμφωνίας και να γίνει διεύρυνσή της γιατί από τότε έχουμε πιο σύγχρονες συμφωνίες και άρα χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε τον προστατευτισμό και έτσι να βοηθήσουμε στον, ε, στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού. Ε, πρέπει να ανοίξουν οι δημόσιες ε, συμβάσεις κατά πολέμηση της ε, διαφθοράς, βοήθεια στις επιχειρήσεις και για όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις διαβουλεύσεις με την ε, με την κοινωνία των πολιτών και όλα αυτά να περνάνε από την κοινή επιτροπή, την συμβουλευτική. Να υπάρχει ένα κεφάλαιο ε, για τις επενδύσεις ε, αντί των 17 διαφορετικών συμφωνίων που υπάρχουν και θα πρέπει αυτό το σύστημα επενδύσεων να υπόκειται σε πολυμερές ε, δικαστήριο. Επίσης θα πρέπει να προχωρούν υπηρεσίες και στα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχουμε εδώ πέρα ένα κατάλογο ε, που ξεκαθαρίζει ότι εξαιρούνται όλες οι ε, κρατικές δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα όσον αφορά την ε, πνευματική ιδιοκτησία και τις προστατευμένες γεωγραφικέ ενδείξει. Είναι σημαντικό να νομοθετήσουμε όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον για τον πιο σωστό τρόπο για να μπορούμε να έχουμε κάποιες ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες τη δυνατότητα να τις επανακρατικοποιήσουμε. Επίσης όσον αφορά τη συνεργασία στα αριθμιστικά αυτό θα πρέπει να διέπεται από μη υπερχωρητικότητα και θα πρέπει να υπάρχουν τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας και σωστή εφαρμογή των φυτογειονομικών και υγειονομικών αρχών. Επίσης να υπάρχει κάτι για το εμπόριο και για την ε, δυνάμει ε, ανάπτυξη. Και αυτό το σύστημα επίλυση των διαφορών να αφήνει την, ε, το περιθώριο να επιβάλλονται κυρώσεις. Επίσης, κύρωση ε, των όσων προβλέπει ο ΠΟΕ και θα πρέπει να ισχύουν τα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα και ένα κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σαφή στόχο που να αξιολογείται ε, για το εμπόριο και να υπάρχουν κάποια ενεργά μέτρα όπως το ενιαίο παράθυρο. Αυτή η συμφωνία πρέπει να έχει και, ένα κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων, είπαμε. Ε, η Χιλή για πρώτη φορά έβαλε τέτοιο κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις με την Ουρουάη και με τον Καναδά. Πρόκειται για δύο χώρες με διαφορές ε, κυβερνήσεις, μία αριστερή και άλλη φιλελεύθερη και είδαμε ότι αυτό το κεφάλαιο βοηθάει σε κοινωνική ειρήνη. Είναι αποτελεσματικό και εμπορικά. Οπότε σήμερα το πρωί ε, είχαμε το Διεθνές Φόρουμ Εμπορίου και Ισότητας των Φίλων. Και η κυρία Μάλστρομ ανακοίνωσε ότι στη συμφωνία με την Χιλή θα υπάρξει σχετικό κεφάλαιο. Επομένως το κάνουμε μια, τώρα μια καινούργια ιστορική διαδρομή για ένα εμπόριο που δεν έχει αποκλεισμούς και επομένως δεν θα πρέπει η, να μείνει πίσω από τις εξελίξεις η Ευρώπη. Επίσης έκκληση προς Συμβούλιο και προς Επιτροπή για να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις αυτού του Κοινοβουλίου και να μην ξεχνούμε ότι στο τέλος των διαπραγματεύσεων εμείς οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών πρόκειται να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε τη συμφωνία. Και ε, οι συνάδελφοι στην Επιτροπή πρόκειται να είναι στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουν τη βοήθειά τους. Thanks um, Σας ευχαριστώ πολύ. Η Έμα Μακλάρκιν έχει το λόγο εκ μέρου των συντηρητικών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια, ε, με την οποία συμφωνούμε πάρα πολύ. Είναι πράγματι αναγκαία η μεταρρύθμιση και ο εξυγχρονισμός συμφωνίας με την Χιλή, ιδιαίτερα ε, ό,τι αφορά το εμπόριο. Νομίζω πως η συμφωνία αυτή ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για εμάς. Και η Χιλή είναι ένα από τα πιο σταθερά κράτη της ε, Λατινικής Αμερικής. Ήταν λοιπόν ε, μια συμφωνία που οδήγησε σε ε, αυξημένη οικονομική δραστηριότητα. Είναι λοιπόν η Χιλή ένας από τους ε, σημαντικούς εμπορικού εταίρου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται παράλληλα με τι διαπραγματεύσει τη ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Μερκοσούρ, είναι ενδεικτικέ ε, τη καλή σχέση που έχουμε. Ελπίζουμε λοιπόν οι αρχές της πολιτικής, όπως μας παρουσιάστηκαν εδώ, να ε, παραμείνουν και στην, ε, στον εξυγχρονισμό της συμφωνίας. Ωστόσο υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά το, το 1D το κομμάτι όπου αναφέρονται οι διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης. Εδώ νομίζω πως χρειάζεται να αναφερθούν συγκεκριμένα μέτρα ε, και συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, θεωρεί τουλάχιστον η εισηγήτρια. Επίσης χρειάζεται να αναφερθεί κάποια ε, ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία θα ισχύει σε όλη τη συμφωνία. Όταν ζητούμε από τους, Ευρω... από τους εταίρους μας να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, τι φανταζόμαστε να περιέχει αυτή η ρήτρα. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που μας απασχολούν καθώς επίσης και ε, οι διατάξεις εφαρμογή του κεφαλαίου για την βιώσιμη ανάπτυξη, του κεφαλαίου για την επίλυση διαφορών, για τις κυρώσεις. Εδώ στις κυρώσεις έχουμε κάποιες αντιρρήσεις. Όπως ξέρετε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση και αυτή η οριζόντια τακτική που ακολουθείται έχει δημιουργήσει εντάσεις. Είμαστε όμως πολύ θετικά προσκύμενοι, θέλουμε να προχωρήσουμε και να προχωρήσει η συμφωνία, γι' αυτό λοιπόν ε, θα δείξουμε κάθε καλή θέληση συνεργασία με την εισηγήτρια. Νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο υπάρχουν κάποια σχόλια από την Επιτροπή για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμφωνία με την Σιγκαπούρη και τον εξυγχρονισμό αυτής θα ε, ήταν καλό να μάθουμε αν αυτή η, η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να επηρεάσει τη συμφωνία με τη Χιλή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Θα εκ μέρου των ε, φιλελεύθερων το λόγο έχετε εσεί, κύριε Χάντσοφα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς χαιρετίζουμε την ε, συμφωνία με την Χιλή. Όπως ανέφεραν και άλλοι, είναι ένα πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρος τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μια χώρα με την οποία μοιραζόμαστε πολλές ε, αξίες. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε όντως να επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία, τις σχέσεις μας και να τις ε, φέρουμε στο παρόν. Όπως είπε και η συγγήτρια, πρέπει να πασχίσουμε να βελτιωθούν τομείς όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις, οι δημόσιες συμβάσεις, όμως εγώ θα έλεγα πως πρέπει να προχωρήσουμε και πέρα από αυτές και το κεφάλαιο για την ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς και άλλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, θεωρώ πως χρειάζεται και εδώ φιλοδοξία. Η χώρα μου είχε συνάψει συμφωνία με την Χιλή, πρωτού προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν να υπάρχει και ένα αντίστοιχο κεφάλαιο για ε, αμοιβέ επενδύσεις στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής θα καταθέσουμε και ε, τροπολογίες. Η μόνη αμφιβολία μου, το μόνο ερωτηματικό που έχω είναι για το σύστημα κυρώσεων και για την επιβολή αυτών καθώς και για την αναστολή των ε, κυρώσεων έτσι όπως αναγράφεται στο σχέδιο έκθεσης όμως ε, θα υποβάλω όλες τις τροπολογίες γραπτός Σας ευχαριστώ πολύ εδώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος των σκιωδών εισηγητών. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ γρήγορα τα γεγονότα εδώ στην Επιτροπή. Έρχομαι από άλλη επιτροπή, από ακρόαση, για να ακούσω αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα άκουσα. Ελπίζω να μην άρχισα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρουν πολύ αυτά που γίνονται. Διάβασα και τις δύο εκθέσεις της κυρίας Ροντρίγκε και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχάς να πω ότι η συνεργασία ε, είναι άψογη στη, μεταξύ των εσκιωδών και με την κυρία Ροντρίγκε και με τη, τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας για τη Χιλή. Ε, νομίζω πως ο πώς έχουν τώρα τα πράγματα στη Λατινική Αμερική κυριαρχούν ανισότητες. Ανισότητες στην ανάπτυξη, ανισότητες στις ε, αξίες. Με τη Χιλή όμως μοιραζόμαστε πάρα πολλά. Έχουμε πολλές κοινέ αξίες, έχουμε κοινή, ε, κοινό πολιτισμό. Η Χιλή έχει δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002 και έχουν γίνει πάρα πολλά. Ε, έχει έρθει όμως η ώρα να επικαιροποιηθεί η συμφωνία, η οποία είναι αρκετά παλιά πλέον. Πρέπει να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η κυρία Ροντρίγκε είπε κάτι που έτσι μου έκανε πολύ ε, εντύπωση. Είπε ότι και η Χιλία από την πλευρά της έχει δείξει μεγάλη θέληση να ξυγχρονίσει τη συμφωνία. Νομίζω πως πρέπει και εμείς να δείξουμε αντίστοιχη προθυμία, να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες έτσι ώστε η συμφωνία να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερο και να είναι επίκαιρη, να είναι σύγχρονη. Το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετό φιλο, αρκετά φιλόδοξο, όμως βλέπω ότι και σε αυτό το προπαρασκευαστικό στάδιο τα πάμε καλά. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ στενή ανάμεσα στη δική σας επιτροπή και τη δική μου αντιπροσωπή, την της Χιλής έχουμε, έχουμε κοινέ ε, συνεδριάσεις, μια κοινή επιτροπή. Νομίζω πως η συνεργασία μας είναι πάρα με την ε, Χιλή και με την ε, πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό θεωρώ πως μπορούμε να συνοδεύσουμε όλες τις διαπραγματεύσεις και τις συνομιλίες σας επαρκώς. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Έχουμε κρατήσει ανοιχτούς όλους ε, τους δρόμους. Είμαστε δεκτικοί και πρόθυμοι για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία που θα καταργήσει όλες τις ε, διμερείς συμφωνίες που έχουν τα κρατημέλη με την ε, Χίλη. Νομίζω πως θα συνεισφέρουμε σημαντικά στον εξυγχρονισμό του συνόλου της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Αυτό που με χαροποίησε πάρα πολύ στην όλη διαδικασία ανταλλαγή απόψεων είναι η αναφορά στην διαφάνεια. Είναι η απέτηση να βελτιωθεί η διαφάνεια. Το είδα όμως όχι μόνο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την πλευρά της Χιλής. Έχει αυξηθεί η διαφάνεια, έχει αυξηθεί ο διάλογος με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ε, αυτό είναι κάτι καινούργιο, ένας νέος δρόμος για την ε, πολιτική ηγεσία της Χιλής. Είναι πάρα πολύ ανοιχτή, θέλουν να χαράξουν και εκείνοι ένα νέο δρόμο στην εμπορική τους πολιτικής εμπορική τους πολιτικοί έχουν ε, λοιπόν ε, δείξει μεγάλη πρόοδο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ε, είναι τόσο θετική και πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις. Κάτι σχετικά με την συμφωνία τώρα. Συμφωνία για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. στην ε, βιολογική γεωργία, στα βιολογικά προϊόντα, τόσο στη Χιλή όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση ετικετών τόσο στην Χιλή όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αλλάξει πολλά στη Λατινική Αμερική και πιστεύω πως ε, όλο αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τους παραγωγούς στη Λατινική Αμερική, στην Χιλή, καθώς επίσης και για τους καταναλωτές εκεί. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω πως η κυρία Ροντρίγκες ε, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και εύχομαι να προχωρήσει γρήγορα, να πάει στην Ολομέλεια το συντομότερο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα ανοίξει το δρόμο για ε, τον εξυγχρονισμό όλων των αντίστοιχων συμφωνιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να επανέλθω στο αρχικό σας σχόλιο. Η Επιτροπή αυτή πάντα εργάζεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Με ακρίβεια και είναι πάντα προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Ναι, δεν αμφέβαλα ποτέ, κύριε Κρέλ. Ο κύριος Αλαφράγκα έχει το λόγο. Όπως τόνισαν και προλαλήσαντε, η Χιλή είναι υπόδειγμα συνεργασίας μεταξύ Ένωση τρίτης χώρα, μια από τις πρώτες χώρες με την οποία κλείσαμε τέτοια συμφωνία ε, συνεργασία με την Δημοκρατική Ρετρατή τη Γενιά και έχουμε τώρα τέταρτη γενιά με το στοιχείο του ελευθερού εμπορίου και όπως είπε και η κυρία Κρέλ, η επικεφαλής της αντιπροσωπείας, η συγκήτρια και η συμφωνία έφεραν πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα Νομίζω ότι η σημερινή προσπάθεια εξεχρονισμού είναι πολύ σημαντική γιατί το, το επιβάλλει η συγκυρία σε σχέση με το ότι όλα άλλαξαν από την τελευταία συμφωνία και έχουμε την σχετική συμφωνία σύνδεσης συνεργασία και άρα τώρα πάμε για πιο φιλόδοξη συμφωνία, πιο σύγχρονη συμφωνία σύμφωνη με την συγκυρία. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Μάτο και συμφωνώ με την προσέγγιση του. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα εξή τρία τα οποία μας παρουσίαζε η κυρία Πινέρο. Πρώτα-πρώτα να υπάρξει απλούστευση των κανόνων προέλευσης, επίσης ε, ανταλλαγή επενδύσεων και πρόεδρε σίγουρα νομίζω ότι η, ο τομέας των ε, υπηρεσιών δεν έχει ρυθμιστεί εξαντλητικά με την ισχύουσα συμφωνία ξέρω το ότι με φωνή βόντος ε, εν τη γιατί πολλά, πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα δεν συμφωνούν, αλλά είναι το πόσο σημαντικό είναι τώρα ε, ο παράγων χρόνος. Ακούσαμε όλοι τι είπε η Επίτροπος Μάλστρομ στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου για τις προτεραιότητες της, ε, του θεματολογίου μας. Και επομένως είπαμε ότι είμαστε τώρα ε, θα κάνουμε εκλογές στη Χιλή, θα έχουμε και εμείς ε, τώρα την αντίστοιχη μέτρηση για τις επόμενες ευρωεκλογές. Και άρα αυτό είναι ένα χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά που λέει η έκθεση, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να αφαιρόμαστε πατερναλιστικά. Είναι η μικρή χώρα, η χιλή, αλλά μεγάλη όσον αφορά και σπουδαία όσον αφορά τις αρχές που συμμεριζόμαστε. Έχουν προχωρήσει πολύ και είναι πάρα πολύ σωστά αυτά τα οποία αναφέρει η έκθεση για αμοιβαία ωφέλεια. Οπότε, Πρόεδρε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε το χρονοδιάγραμμα της Επιτρόπου. Μπορεί να τηρηθεί και να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και μακάρι να έχει έσει του αυτή τη διαπραγμάτευση που δεν νομίζω ότι φαίνεται να είναι ακαθόδηση. Και επομένως νομίζω ότι χωρίς δυσκολίες πριν το τέλος της θητείας αυτής θα έχει εγκρίνει τη συμφωνία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ματίας Γιώργενσεν από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, γνωστός, και ο κύριος Μάρτιν Πλάσα από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Ε, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Πλάθα ονομάζομαι από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. δεν μπορούσε να παραστεί ο τμήματάρχης μου και τον αντικαθιστώ. Να απαντήσω σε αυτά που λέει ο κύριος Μάτο όσον αφορά ε, τις ανησυχίες για την ε, βιολογική παραγωγή. Τα λέει όλα η έκθεση, τι να προσθέσω. Εξηγήθηκαν όλα. Όλα όσον αφορά τα πλεονεκτήματα αυτής της συμφωνίας. Πάντως, τονίζω ότι με διαφάνεια η Κομισιόν ενημέρωσε και πριν αρχίσει η διαπραγματεύση τον Νοέμβριο του 2015 και τον Μάρτιο του 2016 πριν αρχίσει η διαδικασία μονογράφηση της συμφωνίας. Και ενημερώσαμε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για το πού βρισκόμαστε. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις ανησυχίες που έλεγε ο κύριος Μάτο για την ισοδυναμία, να τον καθησυχάσω και αυτόν και τους ε, γεωργούς για αυτές τις ενεργές ουσίες των τρίτων χωρών όσον αφορά αυτές τις συμφωνίες αντιστοιχίες και αναγνώρισης. Είναι προτεραιότητα αυτά για την γενική μας διεύθυνση και όλες οι ουσίες που χρησιμοποιεί η χιλή τις έχουμε αξιολογήσει και τις ε, εγκρίναμε για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η χιλή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να προσαρμοστεί και σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και κόψανε κάποιες ουσίες που δεν χρησιμοποιούμε εμείς. Άρα υπάρχει τώρα αντιστοιχεία και αμοιβή αναγνώριση. Τώρα, όσον αφορά τους ελεγκτές προς τις τρίτες χώρες, σας λέγω ότι η έκθεση αυτή δεν διαφέρει από τις εκθέσεις της υπηρεσίας για κτηνοτροφικά και διατροφικά θέματα, κτηνιατρικά τέλος πάντων και διατροφικά Ακριβώ όπω λοιπόν και οι ελληνικοί μηχανισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ε, το ενδεχόμενο όταν κάτι βρεθεί ω παρατυπία ε, επισημαίνεται και λαμβάνονται μέτρα. Και αν δεν από την τρίτη χώρα, τότε λαμβάνουμε μέτρα Εμεί. στην Ινδία, ω παράδειγμα, εκεί δεν υπάρχει εμβία αναγνώριση για κάποια μεταποιημένα προϊόντα. Ε, και nada más por mi parte. Muchas gracias a todos. Buenas Αυτά και ευχαριστώ. Ματίας. Thank uh, Ο Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια σύντομα σχόλια να κάνω. Είναι εξαιρετική η σχέση με τη Χιλή, όπως είπανε πολλοί. Είναι καλή η συμφωνία μας, αλλά έχει περάσει καιρός. Και όλα πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν, να εξυγχρονιστούν. Οπότε θέλουμε να υπάρξει φιλόδοξο, φιλόδοξο εξυγχρονισμός ε, της ε, συμφωνίας, να αλλάξουμε άρδιν κάποια τμήματα. Τι σημαίνει αυτό? σημαίνει ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα στη φορά την πρόσβαση στην αγορά, τις υπηρεσίες, τα αγαθά, τις δημόσιες προμήθειες. Θέλουμε καλύτερους κανόνες σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τις γεωγραφικές ενδείξεις. Θέλουμε να αντικατοπτρίζει την ε, νέα κατάσταση ε, η συμφωνία και την προστασία και την στήριξη των ε, επενδύσεων και θέλουμε να αντικατοπτρίζεται αυτό που είπαν και αρκετά ε, μέλη της Επιτροπής σας, ότι ε, πρέπει να ε, σεβαστούμε την ατζέντα που έχουμε και θέλουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας και σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά το, το εμπορικό θεματολόγιο όπως υπόθηκε και στη σημερινή διάσκεψη. Τώρα, για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το σχέδιο ψηφίσματος έχει υψηλό επίπεδο ε, φιλοδοξίας, τονίζει και τα θέματα της εφαρμογής. Για την εφαρμογή γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και πρέπει να μελετήσουμε και το αποτέλεσμα του αποτελέσματος της ε, διαβούλευσης της Κομισιόν για την εφαρμογή που έχει ξεκινήσει και με την οποία θα προχωρήσουμε με το Κοινοβούλιο και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Για την βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν και το εμπόριο, να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Το σχέδιο ψηφίσματος ζητά την κύρωση και την άμεση εφαρμογή κάποιων ε, συμβάσεων τις οποίες ωστόσο δεν έχουν κυρώσει όλα τα κράτη-μέλη. Και το λέω αυτό γιατί συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων για την ε, αποτελεσματική εφαρμογή αυτή της ε, συμφωνία, θα μπορούσε να σημάνει ε, υποχρέωση για τα κράτη-μέλη που δεν την έχουν κυρώσει να την κυρώσουν. Αλλά γενικώ είμαστε πολύ θετικοί ε, απέναντι σε αυτό το ψήφισμα, το σχέδιο ψηφίσματος. όντω έχει υψηλό επίπεδο ε, ε, φιλοδοξίας και θεωρούμε ότι θα είναι πολύ χρήσιμο και για εσά. και βεβαίω έχει, χαιρόμαστε που έχει α, ε, τύχει τόσο θετική ανταπόκριση από εσά σε ό,τι αφορά τη χείλη. Ευχαριστώ. Για το θέμα της εφαρμογής και τα εργασιακά κεφάλαια, θα επαναλάβω τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς στις 10 Μαΐου. Είπε θα χρειαστεί όλες οι συμφωνίες οι να συμπεριλαμβάνουν δεσμευτικές ρήτρε για κοινωνικά θέματα και εργασιακά και ε, εισάγοντας ε, εμπορικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των ρητρών. Οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρα τα πράγματα σε ό,τι φορά τη θέση της Επιτροπής για αυτές τις συμφωνίες. Να ακούσουμε τώρα την εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συζητητές και την ε, πρόεδρο της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη δουλειά τους, για την υποστήριξή τους που ανέκαθεν μας πρόσφεραν. Επισημαίνω ότι είναι αλήθεια. Είναι φιλόδοξη αυτή η συμφωνία. Αλλά υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες προς τούτο. Όλοι ενδιαφερόμαστε να είναι μια τέτοια αυτή η συμφωνία και η Χιλή όχι μόνο σε μια ίδιες αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επιπλέον μας, για να μας δημιουργεί εμπιστοσύνη, γιατί κάνουν αυτά που σκέπτονται. Υπάρχει εμπιστοσύνη επομένω σε διαπραγματευτές και σε κυβέρνηση. Και έτσι μπορούμε να βαδισουμε χερι χέρι-χέρι. Οπότε τώρα ε, είδατε τι γίνεται στη διεθνή σκηνή, τι απειλές επικρέμονται να, ένα μήνυμα να στείλουμε στον κόσμο, ένα μήνυμα αισιοδοξία. Όλοι προς αυτό θα προχωρήσουμε. Συμφωνία, φιλόδοξη, με κεφάλαιο για βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αναφέρθηκε, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος Τίμερμαντς, θα πρέπει να έχουμε ένα κεφάλαιο δεσμευτικό για τα κοινωνικά, για τα δρόμενα δικαιώματα. Και θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό που υπογράφουμε και εμείς και η χιλιανοί θα το κάνουμε. Οπότε θα είναι αυτή η συμφωνία σημείο αναφοράς. Γιατί ο κόσμος θα δει ότι καλύπτουμε τον μισό κόσμο. Τις γυναίκες μια βάζουν αυτό το κεφάλαιο για την ισότητα. Έτσι θα είναι. Και θα γίνει αυτό με συνεργασία όλων. 22 έκτου είναι η προθεσμία στις 6 η ώρα το απόγευμα για τις τροπολογίες. Και 11 εβδόμου πρόκειται να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Άρα, ω συνήθω διεκπεριώνουμε ταχαίω. Κύριε Σαλβράνκα, είδατε, όπως είπατε κι εσεί. γρήγορη διαδικασία κύρωσης. Και τώρα... Πάμε στην σύντομη μας ακρόαση για τα δικαιώματα Η ιδιοκτησίας στο σημείο 26 της σημερινής διάταξης. So. Um, λοιπόν, φτάσαμε στη σύντομη μας ακρόαση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχουμε καλέσει δύο εκλεκτούς προσεκτημένους, τον Αντώνιο Καμπίνο, εκτελεστικό διευθυντή της, ε, του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς ήλθατε. Και τον Κάρλος Κορέα, καθηγητή στο κέντρο δια... διεπιστημονικών σπουδών για πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, οικονομικά, νομικά. Έχουμε και βιντεοδιάσκεψη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει το τεχνικό τμήμα εάν μπορούμε να κάνουμε τη βιντεοδιάσκεψη. Ναι, υπέροχα. Τέλεια. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καινοτομία εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βελτιωθούν οι εισαγωγές και ως εκ τούτου να διασφαλιστούν θέσεις απασχόλησης στη βιομηχανία μας. Η Συμφωνία TRIPS αποτελεί το παγκόσμιο πλαίσιο με κανόνες παγκοσμίως Και στις διμερείς συμφωνίε Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε και αρκετέ διατάξει σχετικά με τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, όπως για παράδειγμα στη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Φυσικά, εδώ το ερώτημα είναι εάν αυτό το πλαίσιο είναι επαρκές και αν είναι επαρκές ε, σε παγκόσμια κλίμακα. Προσπαθώντας λοιπόν να αποκτήσουμε μια ευρύτερη εικόνα της κατάστασης με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, διοργανώσαμε αυτήν την ακρόαση και θα αρχίσω με τον πρώτο κύκλο ανταλλαγής απόψεων με τους εμπειρογνώμονές μας και θα δώσω αμέσως το λόγο στον Αντώνιο Καμπίνος. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτήν την ακρόαση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Λάνια για την πρόσκληση η οποία είναι η δεύτερη ε, πρόσκληση. Η πρώτη ε, φορά που βρέθηκα στην Επιτροπή σας ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. Να σας ε, υπενθυμίσω την συνεισφορά της υπηρεσίας μας στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Καταρχάς η υπηρεσία μας προσπαθεί να εναρμονίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την νομοθεσία. Ασχολούμαστε με τα σήματα κατά και τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Είμαστε μια υπηρεσία που λειτουργεί σε άψογη συνεργασία με τα ε, κράτη-μέλη. Περίπου το 70% της ζήτησης ε, για σήματα καταθέντα της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μικρές και μεσαίες. Η υπηρεσία μας χρηματοδοτείται 100% από τους χρήστες μέσω των τελειών που πληρώνουν και με την εξαίρεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που ε, διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρίτες χώρες, οι υπηρεσίες μας είναι ε, δωρεάν, δεν επιβαρύνουν μάλλον τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επίσης αναλαμβάνουμε πλέον αρμοδιότητες όπως ε, συνεργασία, ερευνητικά προγράμματα και σχολούμαστε με θέματα που αφορούν τα την πνευματική ιδιοκτησία ε, συνεργαζόμενη με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Ο στόχος μας είναι να εναρμονιστεί ε, η πνευματική ιδιοκτησία εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό νομίζω πως η παρουσία μας είναι ε, κατάλληλη στη σημερινή ακρόαση. Ο οργανισμός μας είναι ο εκτελεστικός ε, φορέας διαφόρων ε, έργων που χρηματοδοτείται από την Ένωση για την πνευματική ιδιοκτησία σε τρίτες χώρες. Ε, οι διαστηριότητε μα καλύπτουν από την ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της πνευματική ιδιοκτησία στην οικονομία, την κοινωνία και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντα να δημιουργήσουμε καλύτερη κατανόηση των πολιτών για το τι σημαίνει πνευματική ιδιοκτησία. Έχουμε Έχουμε επίσης ε, δραστηριότητες στην Κίνα, την περιοχή ΑΣΕΑΝ, τη Ρωσία και την Ινδία και πρόσφατα υπογράψαμε συμφωνίες ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή τριών ε, project που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στην Κίνα, Νοτιοανατολική Ασία και Λατινική Αμερική. Η χρηματοδότησή μας για αυτά τα τρία project είναι 22 εκατομμύρια ευρώ και οι δράσεις μας διαφέρουν. Έχουμε μία μέση συνεισφορά ε, της τάξης του 15% στον γενικό προπολογισμό του κάθε project προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας πιο αποτελεσματικό για τους χρήστες. Και σε ό,τι αφορά το εμπόριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπηρεσία μας μάλλον, ε, βοηθά τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται παγκοσμίω και να τονώσουν την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα project στόχο έχουν να ενισχύσουν τη την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύσει και την εφαρμογή των συμφωνίων ελεύθερου εμπορίου. Η, η υπηρεσία μας ανέλαβε επιπλέον αρμοδιότητες δεδομένες της σημασίας που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Και γι' αυτό οι αρμοδιότητες ε, που έχει η υπηρεσία μας ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραβιάσεων Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, ενημερώνουμε το κοινό, το ενημερωτικό μας έργο είναι αρκετά σημαντικό και θυμάμαι ότι όταν ο Επίτροπος Μπανιέ μας επισκέφθηκε το 2012 μας είπε ότι σε ό,τι αφορά την παραχάραξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα πρέπει να κατανοήσει τι συμβαίνει και μετά να αναλάβει δράση. Η αποστολή μας ε, έχει διάφορα σκέλη. Καταρχάς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε ε, ουσιαστικά πραγματικά ε, στοιχεία για το πώς ακριβώς συνεισφέρει η πνευματική ιδιοκτησία στην οικονομία και στην ε, κοινωνία του σήμερα. Υπάρχουν έρευνες που έχουν γίνει από την υπηρεσία μας μέσω του παρατηρητηρίου και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών που δείχνει ότι το 38% των θέσεων απασχόλησης, 42% του ΑΕΠ της Ένωσης και το 90% του εξωτερικού εμπορίου ε, σχετίζεται άμεσα με τα δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Είναι λοιπόν άρρηκτα συνδεδεμένη η οικονομία της Ένωσης με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι επενδύσεις που γίνονται το δείχνουν. Επίσης, σήμερα οι τομείς που χρησιμοποιούν την τα πνευματικά δικαιώματα είναι εκείνοι που έχουν τις πιο καλοπληρωμένες θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει και μία έρευνα ε, η οποία εστιάζει στον αντίκτυπο το, της πνευματικής ιδιοκτησίας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Κοιτάζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η έρευνα αυτή αποκαλύπτει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα σήμα κατατεθέν έχουν, είχαν σχεδόν 32% υψηλότερα έσοδα ανά υπάλληλο. Μετά έχουμε δει ότι τα παραποιημένα άγαθα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ένωσης κοστίζουν περίπου 90 δισεκατομμύρια ετησίως και ε, αυτό μεταφράζεται και σε 800.000 θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να το τονίσουμε αυτό. Όλες οι αναπτυγμένες οικονομίες πρέπει να ε, φροντίσουν έτσι ώστε τα πνευματικά δικαιώματα να γίνονται σεβαστά και να υπάρχουν ίση όροι ανταγωνισμού. Τα πνευματικά δικαιώματα που έχουν ένα σταθερό στεγανό πλαίσιο και χαρτίζονται από υψηλή ε, ποιότητα είναι η ελπίδα του μέλλοντος και για τις αναπτυσσόμενες χώρες όμως επειδή ακριβώς θα επιτρέψουν να γίνουν επενδύσεις. Είναι λοιπόν ε, επακόλουθο η παραβιάση αυτών των δικαιωμάτων να μην θεωρούνται μόνο ένα πρόβλημα για αυτούς που κατέχουν τα δικαιώματα, αλλά ε, σοβαρή διατάραξη της αγοράς και κάτι που απειλεί την οικονομική ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν έχει ε, γίνει μια έκθεση η οποία προσπαθεί να χαρτογραφήσει την κλίμακα του προβλήματος και δυστυχώς το πόρισμα είναι ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ ψηλά. Η μελέτη έδειξε ότι ε, σε παγκόσμιο επίπεδο 461 δισεκατομμύρια δολάρια ε, είναι το κέρδος από την πώληση παραποιημένων αγαθών. Το... Και με την ισοτιμία του 2013 αυτό αντιστοιχεί σε 338 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, για να σας το πω και ε, με άλλους όρους, αυτό είναι το ε, συνολικό ΕΠ της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Αυτά τα αντικείμενα που αποτελούν προϊόντα παραποίησης ή πειρατείας αποτελούν το 2,5% του παγκοσμίου εμπορίου και το 5% των εισαγωγών στην Ένωση. Οι ανεπτυγμένες χώρες είναι αυτές που πλήττονται πιο ισχυρά από αυτό το πρόβλημα και βλέπουμε ότι ε, τόσο πρέπει όσο και η πειρατεία ε, ε, αυξάνονται. Αυτά τα φαινόμενα είναι μια πραγματικά παγκόσμια οικονομική απειλή και πολλές φορές συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση εγκληματικών δικτύων που ασχολούνται επίσης με διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση ανθρώπων. Νομίζω έχει έρθει η ώρα λοιπόν να δοθούν λύσεις, να γίνουν δράσεις. Οι χρήστες, οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων το απαιτούν και σίγουρα η λύση δεν μπορεί να δοθεί από μία μόνο ε, πηγή. Δεν μπορεί μόνο ένας οργανισμός να ε, αναλάβει δράση. Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια και ε, ας δούμε ποιοι είναι οι πιθανοί τομεί όπου μπορεί να γίνει αυτή η δράση. Καταρχάς εντό Ένωση. Οι χρήστε ζητούν να γίνουν ε, αναθεωρήσεις, μεταρρυθμίσεις στην οδηγία IP-RED έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερο συντονισμός ε, και εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών. Ζητούν επίσης ε, μία νέα οδηγία για σχεδιασμό και ένα νέο κανονισμό για τον σχεδιασμό, ο οποίος θα είναι ε, ωφέλιμος για την βιομηχανία και για την ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης. Έχει, έχουν δεχτεί με ενθουσιασμό αυτήν την πρόταση όλοι οι φορείς και μάλιστα ε, τον περασμένο Νοέμβριο στο Μιλάνο, στο συνέδριο του Design ε, Europe και υπήρχε σχετική βράβευση. Πέρα από τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζεται επίσης να προστατευτούν όχι μόνο τα οι γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις, αλλά και οι μη γεωργικές, διότι αν δεν βελτιωθεί η νομοθεσία μας, κινδυνεύουμε. Τέλος, ε, πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τη γνώση που έχουμε από ε, τις ε, βιομηχανίες που χρησιμοποιούν έντονα τα πνευματικά δικαιώματα για να καταπολεμήσει το πρόβλημα της ε, ποιητής και της παραποίησης και να συμβάλλει στην ανάπτυξη, την απασχόληση και το εμπόριο. η, ε, η παραποίηση αγαθών είναι κάτι που επίπτει στην αρμοδιότητα του ΠΟΕ και ε, συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συμφωνίας ε, TRIPS. Γνωρίζουμε από μελέτες που έχουν διεξαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι εταιρείε που δεν σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, κοστίζουν θέσεις απασχόλησης από νόμιμες επιχειρήσεις, δεν πληρώνουν φόρους, δεν συμπεριλαμβάνονται στη στατιστικά στοιχεία για την ανάπτυξη. Και επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για μελέτες ε, που χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία και συνεισφέρουν ε, στην οικονομική ανάλυση. ανάλυση. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις για τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ε, το Μεξικό, η Τουρκία, οι 10 χώρες Ασιαν, το Περού και το Μαρόκο. Και νομίζω πως αν καταλάβουμε ακριβώς ε, πώς λειτουργούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την ε, περίπτωση, θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια στρατηγική δράση. Χρειάζεται επιτέλους να ε, ξυπνήσουμε. Πρέπει να δράσουμε για να σταματήσουμε ε, την απώλεια εσόδων για τις κυβερνήσεις, την απώλεια ευκαιριών για ανάπτυξη και την απώλεια θέσεων απασχόλησης που μπορούν να δώσουν ένα, προ, ένα τέλος στην ανασφάλεια για την ανεργία των νέων. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τα πνευματικά δικαιώματα και αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Έχει έρθει η ώρα να αναλάβουμε δράση προς όφελος των ε, πολιτών και των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος, ε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καμπίνος για αυτήν την πολύ περιεκτική παρουσίαση. Τώρα, ελπίζω να μας ακούτε, κύριε καθηγητά Κορέα. Μπορείτε, μας ακούτε, ναι, σας ακούω. Okay. Good afternoon, can you hear me? Good afternoon. So, uh, we will have you uh, on air here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 Έχω την εντύπωση πως τον χάσαμε. Η ψηφιοποίηση του συστήματος ε, δεν είναι τόσο καλή όσο θα περιμέναμε. Γεια σας, ναι, σας χάσαμε. Είμαστε εδώ πάλι. No, we can't hear you. Okay, can you hear me now? That's better. Should I go on?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 Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, για την ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ναι, καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει αυτά που αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε, αλλά το δουλεύουμε. Υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Η κυρία Χάουταλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε η παρουσίαση που μόλις ε, είδαμε από τον Buenos Aires, ομολογώ. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την ευελιξία και τις δυνατότητες που μας δίνει η Συμφωνία Τρίφ στα πλαίσια του ΠΟΕ. Μας είπατε την άποψη το Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να έχουμε καλύτερο συντονισμό έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ευελιξία στα πλαίσια της Συμφωνίας Τρίψ. Η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση. Θεωρείτε ότι αυτός ο προστατευτισμός ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας από κάποιες χώρες ε, θα ε, γίνει σύντομα παρελθόν θα θεωρηθεί παροχημένος ε, όταν συναυτούν αυτές οι συμφωνίες θα υπάρχει ελεύθερη ροή της πληροφορίας. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό θα είναι παροχημένο πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλα σχόλια ή ερωτήσεις. Όχι. Θα δώσω λοιπόν ε, το λόγο πίσω στους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ε, Χάιντι. Ναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ε, θα δεχτώ απαντήσεις και από άλλους συναδέλφους. Όχι, δεν είναι απαραίτητα μια ερώτηση προς τον κύριο Κορέα. Όποιος θέλει να απαντήσει, παρακαλώ να το κάνει. Ναι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει κάποιο σχόλιο από εσά, κάποια ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, ε, αν μου επιτρέπετε, είμαι από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, το τμήμα Άγκρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα στηρίζει την ε, δήλωση της ΔΟΧΑ και στηρίζει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου για αυτό. Η παρουσίαση που μόλις ακούσαμε με μπέρδεψε κάπως, να το <coughs> πω έτσι. Ε, πρώτα αναφέρθηκαν τα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών και μετά ε, συνδέθηκε αυτό με, την, ε, με τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τα προβλήματα αυτά. Ε, υπάρχει ε, διαφορά. Σίγουρα είναι εξίσου σημαντικές όλες οι συμφωνίες, είναι εξίσου σημαντικοί όλοι οι εταίροι μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει αυτή η διευκρίνηση. Μετά για τεχνικά θέματα αναφερθήκε ότι εμείς ζητούμε για προστασία των δεδομένων στα, ε, στις ε, ιατρικές ε, δοκιμές, φαρμακευτικές δοκιμές στα πλαίσια της συμφωνίας TRIPS. Αυτή τη στιγμή έχουμε παγιώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας TRIPS. Υπάρχει προστασία 20 ετών για τις πατέντες. Εδώ έγινε λόγο μόνο για τα φαρμακευτικά και τα χειρουργικά προϊόντα, αλλά ο κατάλογο είναι μακρύ. Χρειάζεται να προστατευτούν οι καταναλωτέ και το κοινό και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη εγγυόμαστε προστασία τουλάχιστον 5 ετών. Αυτή η ειδική προστασία ισχύει μόνο για τέτοιες περιπτώσεις και μπορεί να αυξηθεί στο μέγιστο ε, για 15 χρόνια. Δεν ξεπερνά τα 20 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος λοιπόν πίσω στους εμπειρογνώμονες. Κύριε Καμπίνος, δεν έχετε κάποιο σχόλιο. Κύριε Κορέα. In what I get through internet. But I've heard the, uh, the representative of the European Commission saying that uh, there are no free trade agreements entered into with uh, developing countries.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 and also with Tunisia. So I cannot understand how it it is possible to state that there is no problem with developing countries with agreements which are entered into with the European Commission. Go back to the Commission. Talking about at least... ε, ο λόγος πίσω στην Επιτροπή. Ναι, έγινε λόγος για τα λιγότερα αναπτυγμένα κράτη που ε, καλύπτονται από την ε, διακήρυξη της Ντόχα. Μάλιστα. Ωραία. Χάιντι, έχει το λόγο. Δεν νομίζω πως έλαβα απάντηση από τον κύριο Κορέα. Δεν ξέρω αν ήμουν Ε, Κύριε καθηγητά, κύριε Κορέα, μπορείτε να απαντήσετε στην κυρία Χαουταλά. Well, you know, it was not, I, I couldn't really get the question huh, because uh, there was a problem, problem with the system. I, I started to, uh, to get the question about how to increase uh, the coherence within Europe regarding the policy in order to respect flexibilities for in the area of the in in the area of public health. But I don't know whether this was the question really. Perhaps Heidi, you can raise it again. Heidi, μήπως θα μπορούσες να κάνεις την ερώτησή σου ξανά. Ναι, ας μην αφήσουμε την τεχνολογία να μας ε, χαλάσει αυτή την ωραία ευκαιρία που έχουμε. Θα επαναλάβω λοιπόν. Ε, μιλήσατε για την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Κορέα. Είπατε πω ζητούμε από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις ευελιξίες που δίνει η Συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ και να ποσοτικοποιήσει και να διευκρινίσει ε, όπου χρειάζεται τι συμβαίνει. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις από εσά, Πού μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ποιε είναι οι ευκαιρίε που έχουμε. Και έπειτα, Εσείς θεωρείτε ότι αυτός ο προστατευτισμός στα πνευματικά δικαιώματα που βλέπουμε στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου είναι κάτι το παροχημένο, δηλαδή θεωρείτε πως όλα θα πρέπει, δηλαδή εννοώ το ότι όλα πρέπει να ρέουν ελεύθερα εκτός από τη γνώση, εκτός από ε, αυτό. Yeah, I, I think that there is a clear contradiction between what is being uh, said by the European Commission and the communication I refer to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 Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Α, συγγνώμη, ο κύριο Ντάρτμουθ. Μια που έχουμε χρόνο, ή εκτό αν δεν έχουμε χρόνο, πείτε μου, πρόεδρε. Είναι πραγματικά συναρπαστική η συζήτηση αυτή. Και πρέπει να συγχαρώ τον συνάδελφο που κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Βεβαίω θα πρέπει να. Το πρόβλημα δεν είναι να ακούσουμε τα σχόλια του πάνελ, αλλά αν κάποιο κάτι εφεύρει θα πρέπει να μπορεί να υποφεληθεί από αυτό που εφήβρε. Χωρίς να του πάρουν τα πάντα. Yeah, because somebody invents some medicine. Η... Βεβαίως τα φάρμακα πάντα είναι πολύ πιο δύσκολο να τα εφεύρει κανείς. Ε, ε, ένας με, μικρο... με μικροσκόπιο κατάφερε να βρει την να εφεύρει την πενικυλίνη, αλλά Ουσιαστικά γίνεται κοινό, κοινό κτήμα χωρίς να υπάρχει έξτρα κόστος και κανείς δεν παίρνει κάτι πίσω από την ε, επένδυσή του, άρα υπάρχει πρόσκομα στο να εφεύρει κανείς νέα φάρμακα. Βέβαια, εγώ έχω διάφορες απόψεις και ο πρόεδρος, ο πρόεδρος εδώ και ένα μισή χρόνο ανέχεται όλες μου τις απόψεις και δεν ξέρω και ε, τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά ίσως ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ παρόλο που έχω απόψει πολλέ, δεν έχω λύση για αυτό το γρίφο. Ίσως θα πρέπει να απαντηθούν κάποιο τέτοιο είδους ερωτήματα. reaction of the panelists? Έχετε κάτι να πείτε? This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 Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο πάνελ των ομιλητών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Κομισιόν πρέπει να ακούει περισσότερο το Κοινοβούλιο. Εμάς απολύτως μας ικανοποιεί το μήνυμα αυτό. Και πάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Έχουμε άλλους δύο εμπειρογνώμονες, την κυρία Μαρή Πατούγιο manager στην AIM, European Brands Association, καλώς ήρθατε, και τον Πιότρ Στρεσόφσκι. From the OCD. So uh, now we switch a little bit to the economic and industry. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα την πιο οικονομική διάσταση των πραγμάτων και να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Μαρή Πατούγιο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ξεκινήσω ε, λέγοντας ότι δουλεύω στην προστασία των εμπορικών σημάτων. Ευχαριστώ να μπω και σε θέματα ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά αν μπείτε σε λεπτομέρειες η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου τα ξέρει καλύτερα, σίγουρα. Όπως είπατε, δουλεύω για την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορικών Σημάτων. Ε, σήμερα θα μιλήσω για τη βιομηχανική πτυχή για να σας ε, πω γιατί η AIM εκπροσωπεί 800 ε, περίπου εταιρείε. Ελπίζουμε ότι θα σημαίνουν κάτι όλα αυτά τα εμπορικά σήματα που βλέπετε. Είναι όλα μεγάλη όμιλη προϊόντων. Και Έχουμε, βλέπετε, τη γεωγραφική κάλυψη μέσα των εθνικών ενώσεων. Ε, ελπίζω ότι δεν έχω παραλείψει κάποιον που έρχεται από χώρα που δεν είναι με μπλε χρώμα. Ε, απλώς είναι ότι δεν έχουμε εκεί εθνική ε, εκπροσώπηση. Δουλεύω λοιπόν στα εμπορικά σήματα και στην αντιμετώπιση της παραχάραξης. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες επιτροπές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και εγώ θα επικεντρωθώ στη δεύτερη γιατί η ε, Επιτροπή αυτή για την αντιμετώπιση της παραχάραξης είναι ε, μια, ένας συνασπισμός. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε τόσο εκεί, αν μπορείτε όντως να μου πείτε ποιος είναι ο οπτικός σας γιατί κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι λοιπόν, ε, έχουμε πάρα πολλούς ομίλους εταιριών, ε, τομεακές ενώσεις, ε, παγκόσμιες, εθνικές, ομάδες που δουλεύουν σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση παραχάριξης, όλες με σκοπό να αντιμετωπίσουν αυτήν την απειλή των, της παραχάραξης. Τι γίνεται τώρα με την προστασία των εμπορικών σωμάτων, γιατί υπάρχει. Αφήνοντα όλα τα νομικά στοιχεία, ένα ε, εμπορικό σήμα είναι ένα σήμα καταγωγή ουσιαστικά για τον καταναλωτή. Πάμε σε ένα μαγαζί, βλέπουμε το εμπορικό σήμα, ξέρουμε ότι μπορούμε να το εμπιστευτούμε, γιατί πάνω σε αυτό βασίζεται η, ε, η εταιρεία πάνω στην οποία, ή ε, από την οποία θέλουμε να α, καταναλώσουμε. Είναι λοιπόν ένα, μια συμφωνία εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή. Και έτσι πάμε στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα, γενικώ στην ανάπτυξη και βεβαίω στην ενίσχυση της απασχόλησης. Έχει σημασία η παραχάραξη. Έχω 15 χρόνια που το λέω ε, ότι αν κάποιος μπορεί να το φτιάξει, κάποιος σίγουρα μπορεί να το παραχαράξει. Στην δική μου την υπηρεσία Έχω ε, ψεύτικες τσίχλες, έχω ψεύτικη κρέμα σώματος, έχω παραχαραγμένα ε, προϊόντα διαφόρων ειδών. Μπορεί κανείς να βγάλει πάρα πολλά παράνομα χρήματα με αυτή την, από αυτή την βιομηχανία και είναι βεβαίως απάτη απέναντι στον καταναλωτή. Μπορείτε να νομίζετε ότι ξέρετε ε, αγοράζετε ένα παραχραγμένο προϊόν γιατί είναι πολύ φθηνό ενώ είναι προϊόν μάρκας αλλά δεν έχετε ποτέ ιδέα τι ακριβώς θα πάρετε στα χέρια σας τελικά. Αν αγοράσετε σαμπουάν ή κρέμα σώματος ή κάτι, ένα αντιλιακό έχει την ίδια τιμή με το, με το πραγματικό προϊόν ε, αλλά δυστυχώς δεν σας προσφέρει την ίδια προστασία με το πραγματικό προϊόν. Ακούσατε από τον εκτελεστικό μας διευθυντή κάποια στοιχεία αριθμητικά και είπε ότι στις τομεακές ε, μελέτες βλέπετε ακριβώς πόσο κοστίζει τελικά και σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και, σε το, και στα χαμένα έσοδα. Μιλάμε για 800.000 θέσεις που χάνονται την τελευταία περίοδο. Για τις Βρυξέλλες ας πούμε. 439.705 θέσεις εργασίας στην τελευταία περίοδο αναφοράς. Δύο φορές δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν στην ε, πόλη αυτή έχασαν ε, τη δουλειά τους ακριβώς λόγω της παραχάραξης. Ε, έχει λοιπόν σημασία, φυσικά και έχει. 90 δις χαμένες πωλήσει. Και βέβαια πολλοί, πολλοί λένε «Α, οι καημένες οι πολυεθνικές έχασαν από τα λεφτά τους». Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τα λεφτά τους που πάει να πει ότι απέλεσαν την πολύ κόσμο και αυτό έχει σημασία. Έσοδα από τα φορολογικά. 14,6 ε, δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα. Τον καιρό της λιτότητας δεν νομίζω ότι μπορούμε να ε, χάνουμε 14 δισεκατομμύρια. Και επίσης αυτά τα χρήματα που πάνε. Πάνε σε κάποιον ανταγωνιστή, πάνε σε κάποιον που θα πληρώσει τελικά το προσωπικό του και θα χτίσει ένα ε, εργοστάσιο πάει στο οργανωμένο έγκλημα όπως σας είπαν οι κύριοι εδώ. Είναι, πάνε, πάει στους κακούς της ιστορίας. Ε, έχουμε κάποια στοιχεία και από τους Γάλλους συναδέλφους. Ε, δεν προσπαθώ να ε, σας δώσω ιστορίες από φυλάδες κίτρινες, αλλά είναι πραγματικά δεδομένα αυτά που υπάρχουν από συγκεκριμένες μελέτες. Έχει λοιπόν σημασία? Νομίζω ότι έχει. Τελευταία αριθμητικά στοιχεία για το εμπόριο. 5% των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραχραγμένα προϊόντα. Μόνο ε, εισαγωγές. Δεν μιλάμε για τα πράγματα που κατασκευάζονται εδώ ή που ε, συναρμολογούνται εδώ ή που εξάγονται από εδώ. Είναι αυτά που βρήκαμε εδώ. 5%. Δείτε εδώ γύρω-γύρω στην αίθουσα ένα ε, προϊόν κάθε 20. Είναι παραχραγμένο. Έχουμε μικρά πακέτα, ας πούμε, που έρχονται με το ταχυδρομείο ή με courier και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ελέγξουμε. 5% των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έρχονται όμως μέσω φακέλων, έρχονται σε μεγάλα πλοία, πολύ μεγάλα πλοία. Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση πλοίων ε, εμπορικών. Βλέπετε τον χάρτη. Θα σας πει ο συνάδελφο και άλλα ε, αριθμητικά στοιχεία βέβαια, αλλά 2,5% του παγκοσμίου εμπορίου, δηλαδή 461 δις ε, ε, δολάρια, είναι το 5%. Μιλάμε για τεράστια βιομηχανία. Και 50% όλων των εισαγωγών των προϊόντων που φτάνουν στην Ένωση φτάνουν μέσω μεγάλων πλοίων. Και πού φτάνουν και πάλι δεν μπορείτε να τα δείτε τα στοιχεία αυτά, αλλά πάνω πάνω λέει Ρότερνταμ και το δεύτερο λέει Αμβέρσα. Εξαιρετικά λιμάνια, αλλά δεν είναι οι μεγαλύτερες ε, ε, πρωτεύουσες κατανάλωσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάνουν όμως εκεί για να πάνε αλλού, για να διαμετακομιστούν κάπου αλλού. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε. Οπότε, βεβαίως πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Ένα, Ε, καταχωρούμε τα εμπορικά μας σήματα. Δεν αγοράζετε ε, το αυτοκίνητό σας και το παίρνετε και το αφήνετε με την πόρτα ανοιχτή έξω από την πόρτα του σπιτιού σας και το, κλειδί στην μηχανή. Λέτε ότι είναι δικό μου το αυτοκίνητο αυτό. Το καταχωρείτε λοιπόν. Σε εθνικό επίπεδο, και εδώ πρέπει να πω ότι δεν, το, καταχωρούμε μόνο ε, στο κράτος μέλος μας, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι πολύ γνωστές για τα πλαστά τους προϊόντα. Αν μπορείτε λοιπόν, καταχωρήστε το εμπορικό σας σήμα εκεί. Γιατί ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι η πρώτη γραμμή άμυνας είναι τα τελωνία, τα σύνορα. Μπορούν να σταματήσουν λοιπόν τα, τα προϊόντα μόνο εκεί αν μπορείτε να έχετε καταχωρημένο εμπορικό σήμα. Καταχωρήστε τα εμπορικά σας σήματα. Είπα για τα ατελονία. Το επόμενο βήμα, μόλις ε, λοιπόν έχετε καταχωρήσει, είναι η ε, αίτηση για δράση όπως λέγεται. Ένα έγγραφο δηλαδή που λέει ότι αυτά είναι τα δικαιώματά μου, αυτό είναι το προϊόν μου, αυτό είναι το, ο αριθμός της καταχώρησης και εδώ είναι το τηλέφωνό μου. Α, μία φορά το χρόνο γίνεται αυτό και καμιά φορά βέβαια πρέπει να πείτε και άλλα στοιχεία στα τελωνία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό, αλλά γιατί το κάνουμε. Τα τελωνία μπορούν να ελέγξουν 1,5% του εμπορίου. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτού που κάνουν είναι πριν την ε, άφηξη των προϊόντων, ε, ανάλυση κινδύνου. Και αυτό γίνεται μέσω των άλλων πληροφοριών που παίρνουν. Ξεκινάει ε, να έρχεται ένα ε, προϊόν σε ένα συγκεκριμένο λιμάνι. Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει μια παρόμοια τάση και αλλού. Αυτό λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι να έχουμε την βάση δεδομένων για την εφαρμογή, Οπότε όλα τα στοιχεία αυτά πάνε στις ε, διοκτικές αρχές κατευθείαν. Μπορούν να τα κατεβάσουν τα τελωνία και η αστυνομία και να έχουν τα στοιχεία από, την, ε, από τον κάτοχο του δικαιώματος όμως ξέρουμε ε, ποιος είναι ο κακός της υπόθεσης και ξέρουμε και θα πάμε κατευθείαν στην αστυνομία. Οπότε από εκεί και πέρα η αστυνομία μετά θα χρησιμοποιήσει και θα διαμοιράσει αυτές τις πληροφορίες όπως μπορεί. Τώρα για τα τελωνία δουλεύουμε επί τόπου και με τις ε, αστυνομικές αρχές, κάνουμε ε, επεμβάσεις και Πάμε εδώ στην ανάγκη συνεργασίας με τις ε, αρχές επιβολής του νόμου. Η Όλαφ είναι η καταλληλότερη υπηρεσία, η Interpol επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η Europol είναι πολύ καλή, με μεγάλη διάθεση για βοήθεια και έχουν πολύ καλές εκστρατείες, με πάρα πολύ καλές πληροφορίες, εύληπτες, ε, προσβάσιμες, μπείτε στην ιστοσελίδα και δείτε. Μετά, Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γενική Διεύθυνση ε, ε, Εμπορίου. Γιατί γίνονται διάλογοι, γίνονται συζητήσει, συγκρίνονται τα στοιχεία. Έρχεται κάποιο και λέει, έχετε κι εσεί πρόβλημα, έχουμε κι εμεί πρόβλημα. Α το λύσουμε μαζί. Ακούσατε από τον ε, εκτελεστικό μα διευθυντή το, διάφορε δυνατότητε δυνατότητες παρέμβασης και βοήθεια, Αλλά εφόσον αυτό υπάρχει μέσα στις συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου, θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα, σημαντικό βήμα, όχι μόνο για μας, αλλά και αυτούς με τους οποίους εμπορευόμαστε και που κατασκευάσουν πράγματα και που έχουν ε, εμπορικά σήματα και που θέλουν να συνεχίσουν να κατασκευάσουν τα προϊόντα τους και να έχουν ε, ε, δουλειές. Οπότε είναι αμφίδρομη η κατάσταση, αλλά χρειάζεται εφαρμογή. Σε κάποιες περιοχές του κόσμου διευκολύνονται, διευκολύνεται το εμπόριο νόμιμα. Υπάρχει λοιπόν διευκόλυνση εμπορίου. Αφήστε λοιπόν την, ε, τις διεκτικές αρχές να μπουν σε αυτές τις ζώνες ελευθεροπορίου και να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα, να ευχαριστήσω την ε, ε Κομισιόν και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια. Κάποιος έφτιαξε αυτό το πλαστό ποτήρι, κάποιος το αγόρασε αυτό το πλαστό ποτήρι. Δεν είναι όμως ο κατασκευαστής ούτε το, το, το, το, το, πρόσωπο α ούτε το πρόσωπο β. Κάποιος πήγε, το μετέφερε το, από το σημείο α το σημείο, στο σημείο β. Μπορεί να είναι οι υπηρεσίες των courier, μπορεί να είναι online, μπορεί να είναι κάποιοι ειδικοί ενδιάμεση. Κά, όλοι αυτοί οι ενδιάμεσοι όμως κάνουν, βγάζουν λεφτά από την οποιαδήποτε μετακίνηση του παράνομου προϊόντος. Γι' αυτό πραγματικά χαίρομαι που το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα στις 15 Ιουνίου υιοθέτησε το ψήφισμα για τις online πλατφόρμες και το κείμενο αυτό λέει μεταξύ άλλων ότι, όλοι οι, ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ενδιάμεσοι που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, λαμβάνοντας ε, ανάλογα και αποτελεσματικά μέτρα. Εδώ το θέμα δεν είναι το θέμα της ευθύνη, είναι το θέμα για τις ε, εταιρείε που ε, κάνουν νόμιμα τις ε, δουλειές τους και θέλουν ε, να συνεχίσουν να, κάνουν, να έχουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κοινή λοιπόν η ευθύνη όλων μας και των χαραστών την πολιτική και της βιομηχανίας και των διευθυντικών αρχών αλλά τελικά καταλήγουμε σε δύο πράγματα. Η οικονομική ανάπτυξη και προστασία των καταναλωτών. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές το μήνυμα για τον οικονομικό αντίκτυπο της παραχάραξης. Και ε, τώρα θα δώσω το λόγο ε, στον ε, μας από τον Όσα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Ο οργανισμός μου έχει έδρα στο Παρίσι, αλλά στην ουσία ε, ασχολούμαστε με στατιστικές. Προσπαθούμε δηλαδή, αναλύοντας δεδομένα, να ε, παρουσιάσουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία που βοηθούν στη χάραξη πολιτικής. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθούμε. Είμαστε ένας ε, δημόσιος οργανισμός που ασχολείται με ε, την δημόσια πολιτική. Θα αρχίσω λοιπόν λέγοντας γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει το πόριο ε, πλαστών αγαθών. Γιατί λοιπόν η ε, υπεύθυνοι πολιτικής πρέπει να ενδιαφέρονται για το εμπόριο αυτό. Ε, νομίζω πως η παρουσίαση που ακούσαμε πλαισίωσε την ε, συνέχεια της ε, συζήτησης. Υπάρχουν τάσεις που έχουν διαπιστωθεί και μπορούμε να δηλήσουμε κάποια αρχικά συμπεράσματα. Ε, υπό τον όρο της πνευματικής ιδιοκτησίας υπάγονται διάφορα. Υπάρχει για παράδειγμα, ο τρόπος που γίνεται η παραγωγή και τα εμπορικά σήματα μας λένε πολλά για τους καταναλωτές και για το ίδιο το προϊόν. Αυτό εδώ είναι εμπορικό σήμα. Είναι δικαίωμά μου να πιστεύω ότι αυτό εδώ το αγαθό έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία με το όνομα Halter. Όταν κάποιο ε, ε, παραχαράσει αυτό και δημιουργεί ένα πλαστό προϊόν, τότε ε, παραπλανεί τον καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμο... Ε, βλέπουμε τη χρησιμότητα των εμπορικών σημάτων των, της πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιατί λοιπόν ε, θα ε, πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό. Τα δεδομένα που έχουμε στον οργανισμό μας δείχνουν ότι ο όγκος των πλαστών αγαθών αυξάνεται. Υπάρχουν και διάφορες μελέτες, και οικονομικές μελέτες και άλλες, που δείχνουν πόσο σημαντικά είναι τα εμπορικά σήματα στο ΑΕΠ. Εγώ προσωπικά θα σας πω τη δική μου ιστορία. Μένω στο Παρίσι, είναι μια υπέροχη πόλη και όταν ερχόμουν με το τρένο στις Βρυξέλλες σκεφτόμουν ε, αν υπάρχει κάτι που να μην περιέχει ένα εμπορικό σήμα. Αν οποιαδήποτε απόφαση που ε, λαμβάνω ε, δεν σχετίζεται με κάποιο εμπορικό σήμα. Από το ψωμί και το κρουασάν που αγοράζω ε, μέχρι το σούπερ μάρκετ, μέχρι όταν πηγαίνω στο Καρφούρ και παίρνω ε, το, το τυρί ε, president, έχει και αυτό εμπορικό σήμα. Όλα συνδέονται με αυτό. Λοιπόν, η αξία των εμπορικών σημάτων μεγαλώνει. Αυτό σημαίνει ότι οι παραχαράκτες έχουν τεράστιες ευκαιρίες εδώ δραστηριότητας. Και η δράση τους καλύπτει πάρα πολλούς τομείς, από είδη πολυτελείας μέχρι μεταφορές ταξίδια. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι τις διαδρομές αυτών των, των αγαθών. Πολλές φορές δεν πηγαίνουν από το σημείο Α στο σημείο Β, αλλά από το σημείο Α στο Β, στο Γ, στο Δ, ξανά στο Α. Και έτσι ε, λοιπόν το made in, αυτή η ετικέτα ε, δεν ε, ισχύει πια. Αυτό εδώ το Blackberry, αυτό το κινητό τηλέφωνο. Για να δημιουργηθεί ε, χρειάστηκε κάποιος να το σκεφτεί, κάποιος να το σχεδιάσει, κάποιος να φτιάξει το κάλυμα, τη θήκη, τα chip υπάρχουν πολλές ε, χώρες λοιπόν που εμπλέκονται στην ε, παραγωγή ενός BlackBerry και πολλές ευκαιρίες λοιπόν για τους, ε, ε για τους παραχαράκτες να δράσουν. Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβουμε δράση αμέσως διότι υπάρχει άμεση σχέση προσφοράς και ζήτησης. Φυσικά και είναι πρόβλημα τα πλαστά προϊόντα. Όμως ε, ο οργανισμός μας, όπως σας είπα, είναι ένας οργανισμός ε, στατιστικολόγων. Αυτό που κάνουμε είναι να αναλύουμε τα στοιχεία, να κάνουμε στατιστικές που βοηθούν ε, τους υπεύθυνους πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι εμείς βασιζόμαστε σε στοιχεία. Αν δεν έχουμε στοιχεία βάζουμε ερωτηματικό. Οι μελέτες αυτές είναι ε, ξεκάθαρες, είναι χαρακτηρισμένες από απόλυτη διαφάνεια. Στο τέλος κάθε μελέτης βλέπετε τις πηγές μας, βλέπετε ε, ε τι χρησιμοποιήσαμε και ε, όπως ε, σας είπα, είμαστε ένας δημόσιος ε, οργανισμός και να είστε σίγουροι ότι δεν έχουμε λάβει ούτε, ούτε ένα σέντ για από ιδιώτες, από λόμπι για να κάνουμε τις μελέτες μας. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε μία ξεκάθαρη αντικειμενική εικόνα του όγκου της ε, παραποίησης. Θα ήθελα τώρα να σας ε, παρουσιάσω κάποια στοιχεία, κάποιες ε, φωτογραφίες, κάποιες εικόνες. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την κλίμακα, όπως είπε και ο κύριος Καμπίνο, 461 δισεκατομμύρια δολάρια πλαστών αγαθών ε, κυκλοφόρησαν στο εμπόριο το 2013. Αυτό είναι σχεδόν το 2,5% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου. Είναι δύο φορές τα, ε, ο κύκλος εργασιών της Apple κάθε χρόνο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στόχος. Το 5% όλων των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλαστά. Ε, και το 6,5% του εμπορίου ε, αγαθών υψηλής τεχνολογίας είναι επίσης πλαστά. Πριν από λίγες μέρες ε, αρχίσαμε και μια άλλη μελέτη που καλύπτει άλλα προϊόντα, φάρμακα και φαρμακευτικά σκευάσματα. Και 62 δισεκατομμύρια δολάρια σε φαρμακευτικά αγαθά είναι ε, πλαστά. Αυτοί οι ασθενείς λοιπόν που παίρνουν αυτά ε, τα φάρμακα ε, παραπλανώνται και έχουν το δικαίωμα να ε, ξέρουν ότι τα φάρμακα που παίρνουν είναι γνήσια. Τώρα, ποιο είναι το εύρος, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής. Οποιοδήποτε προστατευμένο προϊόν μπορεί να αποτελέσει στόχο για τους ε, παραχαράκτες για παράδειγμα είδη πολυτελείας, αρώματα, ρολόγια, δερματινά είδη, τσάντες, αλλά και ε, μηχανήματα, χημικά, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά, όταν πας σε ένα συνεργείο ε, και πας στο αυτοκίνητό σου θες να πιστεύεις ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι γνήσιο, αλλά ποιος το εγγυάται. Επίσης, καταναλωτικά αγαθά, ε, παιχνίδια, φάρμακα, καλλιντικά, τρόφιμα, τρόφιμα για μωρά. Εγώ έχω ένα μωρό και όποιος ε, έχει ε, μικρό παιδί είναι διατεθειμένος να πληρώσει αρκετά για να ε, πάρει στο παιδί του γνήσια προϊόντα. Και εγώ αυτομάτως είμαι στόχος. Επίσης, τρόφιμα, ε, φράουλες, μπανάνες, κανέλα, καριδέλαιο, όλα αυτά είναι αντικείμενα για τα οποία οι καταναλωτές δέχονται να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Όλοι προτιμούν να πάρουν την μπανάνα που έχει το αυτοκολλητάκι παρά την μπανάνα που δεν το έχει. Αλλά όταν ε, η μπανάνα που δεν έχει το αυτοκολλητάκι της ε, προέλευσης είναι πάρα πολύ φθηνότερη, τότε αυτομάτως ε, γίνεται ε, ανάρπαστη, γίνεται πιο ελκυστική για τον καταναλωτή. Τώρα, ποια είναι η πηγή όλων αυτών των πλαστών αγαθών. Δυστυχώς οι μελέτες μας και η επόμενη μελέτη που θα ξεκινήσει δείχνει ότι είναι οργανωμένη επιχείρηση η, η είναι μια οργανωμένη επιχείρηση που χρησιμοποιεί όλες τις ε, νόμιμε μεθόδους, ηλεκτρονικό εμπόριο, μεταφορές κτλ. Βλέπουμε ότι η πηγή της παραγωγή τέτοιων πλαστών αγαθών είναι η Κίνα, είναι το κέντρο. Ε, ταυτόχρονα όμως οι κόμβοι διακίνηση είναι διάφοροι, υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστημα ακριβώ για να ε, δημιουργηθούν από τη μία διάφορα κέντρα διανομής ε, σε περιοχές όπου δεν επιβάλλεται ο νόμος, όπως ε, στην προκειμένη περίπτωση Χονγκ Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ε, περιοχές στις οποίες χρειάζεται βελτίωση στην εφαρμογή του νόμου. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες τάσεις, συγκεκριμένα μοτίβα ανάλογα την περιοχή, ανάλογα τον κλάδο. Τώρα, ε, στην Ευρώπη βλέπουμε ότι οι οικονομίες όπως της Αλβανίας, Αιγύπτου, το Μαρόκο και της Ουκρανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ε, αναδιανομή ή την διέλευση πλαστών αγαθών ε, που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Επόμενη διαφάνεια, οι στόχοι. Ποιοι είναι οι στόχοι, ποιε είναι οι εταιρείε που πλήττονται περισσότερο. Βλέπουμε ότι είναι εταιρείε ε, από χώρε του ΟΣΑ, Ηνωμένε Πολιτείε, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο. Αυτέ είναι στην κορυφή τη λίστα. Εταιρείε από αυτέ τι χώρε ε, υποφέρουν πραγματικά από, τα, ε, την παραποίηση αγαθών και τα αποτελέσματα. Έχουν τώρα ως εξής, εμείς συνεργαζόμαστε με αυτές τις χώρες και προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Είναι δυνατόν για, και βασισμένοι σε αυτό να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις μας βασίζονται σε ε, απώλεια εισοδήματος, ε, πωλήσεων, ε, διαφυγόντα κέρδη και ε, θέσεις εργασίας, ε, χαμένες θέσεις εργασίας. Εντοπίσαμε ε, επιπτώσεις στη διαφθορά, στην ασφάλεια, την ε, δημόσια υγεία, με πλαστές μπαταρίες, με πλαστά φάρμακα, με πλαστά φυτοφάρμακα και επίσης υπάρχουν μειωμένα κίνητρα από τις εταιρείες να διαθέσουν νέα προϊόντα στην αγορά. Γιατί δηλαδή να μπει στον κόπο να αναπτύξεις ε, μια νέα τεχνολογία, ένα νέο προϊόν, όταν με το που το βγάλεις μια άλλη εταιρεία θα το αντιγράψει με πολύ μικρότερο κόστος και θα ε, σου φάει τη δουλειά. Μετά, τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι δύσκολη μια απάντηση ακριβώς γιατί αυτοί οι παραχαρακτές ε, δρούν παγκόσμια, δεν έχει σύνορα η πρακτική αυτή, δεν υπάγονται σε κανόνες, σε πρότυπα, σε καμία ε, νόμιμη διαδικασία θεμητού εμπορίου. Υπάρχει λοιπόν μία ε, δυσκολία η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί, ιδιαίτερα, για την, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Όπως σα είπα όμω και πριν, όπω ακούσαμε και πριν, πρώτα πρέπει να κατανοήσεις τι συμβαίνει και μετά να αναλάβεις δράση. Ελπίζω λοιπόν να σας έδωσα μία συνοπτική εικόνα του ε, πώς έχουν τα πράγματα και να μην σα κούρασα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Τώρα οι παρατηρήσει των συναδέλφων. Φάιντι. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και εμεί ω καταναλωτέ. Ε, με τις παραποιήσεις νιώθουμε μεγάλη απογοήτευση, μη σας πω παραδείγματα από προσωπική εμπειρία. Οπότε ακούσαμε για το τι χρειάζεται να γίνει. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για το ότι τέτοιους, τέτοιας κλίμακας παραποίηση έχει κάποια σχέση με την εξωχώρια οικονομία που τώρα είναι στο στόχαστρο του Κοινοβουλίου. Ενδιαφέρεται πολύ τώρα το Κοινοβούλιο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή, τα, τα, την οικονομία την εξωχώρια. Και επίσης είδαμε ότι υπάρχουν διάφοροι κόμβοι τέτοιων παρεμένων προϊόντων που είναι στη γειτονιά μας γύρω-γύρω προς Ανατολάς και προς Νότον. Οπότε αυτό θα πρέπει να μπει στο θεματολόγιο της ε, πολιτικής γυθνίασης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βοηθούσε να είχαμε κάποιο είδου ε, συμφωνία, συνεργασία, Φερρυπίν με την Ουκρανία και να μπορεί να επιληφθεί η Eurojust για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την παραποίηση και τη διάβαση των συνόρων από αυτά τα προϊόντα και να υπάρχουν μόνος κάποιοι μηχανισμοί που να μπορούν να ε, παρέμβουν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φερνάντες, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο όμως. Έλεγα πρόεδρε ότι ευχαριστώ και θέλω και να συγχαρώ τους δύο εισηγητές γιατί μας τα είπανε πολύ ξεκάθαρα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και οι δύο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ας μου απαντήσει όποιος θέλει. Το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Μαΐου εγκρίναμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, ούτως ώστε να ληφθούν μέτρα εναρμόνισης των μέτρων ελέγχου, επιθεωρήσεων και κυρώσεων σε επίπεδο τελωνίων για να καταπολεμηθούν οι παραποίησης. Έχουμε την Τελωνική Ένωση, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Μια που με διάφορους μηχανισμούς ε, επιθεωρήσεων και ελέγχων ε, ακόμα υπάρχουν ε, παραθυράκια για να μπουν παραποιημένα προϊόντα. Και με εκείνη την έκθεση πρωτοβουλίες θέλαμε να βρεθούν κάποιοι μηχανισμοί και να έχουμε ουσιαστική εναρμόνιση. Εσείς θεωρείτε ότι πραγματικά χρειάζεται να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την εναρμόνιση. Θα ήταν χρήσιμο μέτρο για να ελαχιστοποιήσουμε το λαθρεμπόριο και πριν τις εναρμόνισης. Αυτό που δεν καταφέραμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετή πλειοψηφία, να έχουμε μια κεντρική υπηρεσία που να ελέγχει τους μηχανισμούς, τα συστήματα που έχουν σχέση με τα τελωνία. Να ελέγχεται δηλαδή το ότι είναι ίδιες οι διαδικασίες, ίδιες οι κυρώσεις, οι ίδιοι οι μηχανισμοί και τα συστήματα επιθεωρήσεων και ελέγχων. Και έτσι να είχαμε αυθεντική εναρμόνιση. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος, και εγώ έχω να πω μια σκέψη μου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Λέει κάποια μελέτη ότι 54% των χρηστών χρησιμοποιούν για τα, προσόν, για τα προϊόντα τους το ίντερνετ. και έχει διπλασιαστεί ο όγκος του Ιντερνετικού εμπορίου. Αυτό τι συνέπειε για το θέμα μας. Δεν έρχονται δηλαδή στη Βαλένθια ή στο Αμβούργο ή στην Αμβέρσα τα κοντέινερς, αλλά η DHL, κάποιος κουρίερ, παραδίδει το πακέτο με τα παραποιημένα. Νομίζω ότι η κατάσταση έτσι μπερδεύεται περισσότερο, ίσως είναι χειρότερη με το ηλεκτρονικό εμπόριο δηλαδή. Πως πρέπει να κάνουμε κάποια προσπάθεια ρύθμισης μέσω του ΠΟΕ. Αλλά πριν μας απαντήσετε, να απευθυνθούμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σύντομη δήλωση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ε, ευκαιρία αυτή. Η Γενική Διεύθυνση για το εμπόριο μέσω των πολυμερών σχέσεων και των ε, συμφωνιών είναι κάτι το... είναι, είναι μέσα, τα μέσα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το τι γίνεται με το software, με τα καλλιτεχνικά έργα κλπ. Όπως είπε και η κυρία Πατούλιο. Και προσπαθούμε να είμαστε φάνταστοι για όλα τα προϊόντα, για τρένα, τηλεπικοινωνίες, ε, μηχανές, για διάφορα προϊόντα που είναι παγκοσμίου φήμης. Να καλύψουμε και κάποιους που επινοούν, κατασκευάζουν φάρμακα εκπληκτικά που γιατρεύουν ασθένειες. Και αυτά τα φάρμακα είναι ακριβά. Όμως, όλα αυτά να μην γίνονται εις βάρος των φτώχων χωρών. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού. Και θα πρέπει να υπάρχει μια βάση κανόνων για να προστατευτεί η πνευματική ε, ιδιοκτησία. Ενεργούμε επί τη βάση των όσων επιτάσσει το Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ανάπτυξη των χρόνων με τις οποίες ε, διαπραγματευόμαστε. Οπότε, ίσως είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι 95% των φαρμάκων που έχουν καταγραφεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν προστατεύονται από ευρεσιτεχνία. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Μόνο 5% έχουν ευρεσιτεχνία. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι καμία λιγότερο αναπτυγμένη χώρα δεν ε, έχει τίποτε κανόνες ε, πνευματικής ιδιοκτησία. Άρα, αυτά τα φάρμακα δεν πάνε σε εκείνες τις χώρες. Αυτό τι σημαίνει, ότι ίσως το πρόγραμμα δεν είναι πνευματική διοκτησία, είναι αλλού. Δεν είναι φραγμός η πνευματική διοκτησία στην αδυναμία των λιγότερο ανεπτυγμένων να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα. Και δεν λέμε για την ε, θεραπεία του καρκίνου, μιλάμε για φάρμακα, για τις στοιχειώδεις, βασικές ασθένειες, κοινέ. Ακολουθούμε επομένω τις νομοδοτήσει του Κοινοβουλίου, τι εξελίξει για το θεματολόγιο της Ντόχα Αυτά και στις διαπραγματεύσεις εμπορικές και η κυρία Πατρούλα το ανεγνώρισε ότι προσπαθούμε να προωθήσουμε το καθεστώς το οποίο εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο. Για καλά νομοθετήματα, ας πούμε, εναρμόνιση, όπως είπατε, για την τελωνία. Έχουμε έναν κανονισμό σχετικά. Είναι ο πιο προοδευτικός, ο πιο σύγχρονος στον κόσμο. Έτσι τα τελωνία μας μπορούν να κατάσχουν, να δημεύσουν ε, εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμυρίων παρανόμων προϊόντων. Προσπαθούμε και με τις ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις. Πριν μια εβδομάδα είχα πάει στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε ένα project αδελφοποίησης με την ε, Ουκρανική κυβέρνηση. Να θέλουμε να βοηθήσουμε και την ε, Ουκρανία να θεσπίσει κάποιους νόμους για να ε, ευθυγραμμιστεί με τα όσα ισχύουν για τα αναπτυξιακά της ΕΖΕΣ. Πάντως, βοηθάει πάρα πολύ με χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Τώρα για το ηλεκτρονικό εμπόριο δύο λόγια. Όντως, αυτό είναι θέμα σημαντικό. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία που προσφέρεται, αλλά μπορεί όπως όλα να τύχει κατάχρηση από κάποιους και από πλευράς δικής μας προσπαθούμε με το πλαίσιο που έχουμε, τους πόρους που έχουμε, προσπαθούμε σκληρά να έχουμε έναν κατάλογο για το τι πρέπει να ελέγχουμε στην αγορά, των ε, πληροφοριών, της βιομηχανίας, για το παρατηρητήριο. Προσπαθούμε να επισημάνουμε σε ποιες αγορές έχουμε πωλήσει παραποιημένων και απομιμήσεων. Κάμε μια εξτρατεία συνειδητοποίησης και ενημέρωσης. Ε, βέβαια, και έχουμε τις συνομιλίες και την πρόοδο του ελληνικού εμπορίου στον ΠΟΕ. Άρα θα πρέπει να βοηθάμε το ηλεκτρικό εμπόριο αν προσέχουμε να μην γίνεται κατάχρησή του. Η κυρία Πατούγιο έχει τώρα τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να προσπαθήσω να σας ε, απαντήσω. Αν δεν απαντήσω είναι γιατί δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Η εγκληματικότητα συνδέεται και η εγκληματικότητα και το κυβερνό έγκλημα με τα παραπημένα και τις απομιμήσεις. Άρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Τώρα, ο Πιότρ ανέφερε τι θέματα υπάρχουν με τα παραποιημένα που γίνονται στην Ένωση από τους κοντινούς μας γειτόνους και άρα ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε μέσω των κυβερνήσεων της χώρας εκείνες και αυτό έχει σχέση με την επόμενη ερώτηση. Τα τελωνία. Δεν είναι κάποιοι που βαριούνται να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, τελωνιακοί όλη τη μέρα απασχίζουν. Κάνουν πάρα πολλά. Και ας μην ε, έχουν το σεβασμό που τους αξίζει. Σε εκείνες τις χώρες πληρώνονται φυσικά λιγότερο. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε τι απαιτούμε να κάνουμε. Θα ήθελα να αυξηθούν οι πόροι υπέρ των τελών παντού. Το επόμενο βήμα τώρα είναι ότι θα θέλαμε να εκπαιδεύονται οι τελωνιακοί στα θέματα πνευματική διοκτησίας. Ε, ψάχνουν, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Ακόμα και το αμπαλάζ και τη συσκευασία μπορούν να καταλάβουν. Οπότε αυτή η ε, αξιωματική πολλές φορές με τις ειδικές τους γνώσεις προάγονται πάνε σε άλλη υπηρεσία αλλά θέλαμε να μείνει στο τελωνίο. Τώρα όσον αφορά την, την κεντροκατευθυνόμενη ε, διαχείριση έχουμε στην Ευρώπη την Europol που δεν είναι, είναι και αστυνομία, δεν είναι μόνο τελωνία και όπως είπε ο Πέδρο από πλευρά διαδικαστική έχουμε τον κανονισμό που ορίζει τα τελωνιακά, αλλά έχουμε και την ε, σχετική οδηγία. Σε κάποιες χώρε αυτή έχει αποτελέσει ποινικό δίκαιο, οπότε ελπίζουμε ότι θα επικαιροποιηθεί και αυτή η οδηγία. Εσείς το 2004 δώσατε αγώνα για να εγκριθεί αυτή η οδηγία. Μπράβο αλλά θα πρέπει να ισχύσουν καλύτερες, πιο αποτελεσματικές κυρώσεις. Να εφαρμοστεί ο νόμος ως έχει. Επίσης, δεν θα γίνει με τους πόρου μας, όπως είπατε και πριν για το ηλεκτρικό εμπόριο. Όντως έχουμε δέματα κατά εκατομμύρια. Και Πρόκειται για παγκόσμιο εμπόριο, υπάρχουν πολλές δυσκολίε για να βρεθούν, να επισημανθούν, να κατασκευθούν. Ε, τι θα γίνει, θα υποφέρουν περισσότεροι, ναι. Και θα κυκλοφορούν ακόμα διάφορα παραποιημένα ε, εμπόρια. Ε, συγγνώμη, φάρμακα στην αγορά. Και αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός βρίσκεται η λύση. Ποιο τρέχει το λόγο. Θα ήθελα κι εγώ να προσθέσω κάτι, αλλά μπορώ να πω μόνο ότι είναι βασισμένο σε στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τι οικονομίε offshore και τι οικονομίες γύρω από αυτές, οι πληροφορίες μας και οι αναλύσεις μας δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές ζώνες ελεύθερου εμπορίου οι οποίες είναι αντικείμενο κατάχρηση και χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση πλαστών αγαθών ε, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και σε ό,τι αφορά τα εμπορευματοκιβώτια που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι φτάνουν σε αυτές τις ε, ζώνες ελεύθερου εμπορίου, μετά ξεφορτώνονται, φορτώνονται σε μικρότερα δέματα και αυτά φτάνουν με τη σειρά τους μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ε, αυτή η διαδικασία ανασυσκευασίας, αυτή που μειώνει το ρίσκο να σε πιάσουν στα σύνορα. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με τον ε, ΠΟΕΚ έχουμε ξεκινήσει ένα ε, έργο παρακολούθησης που προσπαθούμε να δούμε αυτά ακριβώς τα κέντρα, τους κόμβους εμ, διακίνησης αγαθών και να εντοπίσουμε ποια είναι τα και να ποιες είναι οι ελλείψεις στην διακυβέρνηση, τι κοινωνικές συνθήκες που ευνοούν την ε, ανάπτυξη αυτών των, ε, με, των ε, τοποθεσίων ως Το Χονγκ και, και η Σιγκαπούρη είναι αναπτυγμένες οικονομίες που ωστόσο φιλοξενούν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Η ερώτηση τώρα για την Τελωνιακή Ένωση. Να σας πω ότι υπάρχουν κάποια κενά διακυβέρνησης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν από εσάς μάλιστα έτσι ώστε να ε, επιλύσουμε το πρόβλημα, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Κυρώσεις και ποινές. Οι φιλοσοφοί είναι πάρα πολύ έξυπνοι, είναι καλοί επιχειρηματίες και ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα αδύνατα σημεία και πού να κρυφτούν. Και ε, τέλος για το ηλεκτρονικό εμπόριο να πω ότι είναι εκπληκτική λύση. Το, λατρεύω το Amazon, η γυναίκα μου ψωνίζει από το Ζαλάντο και ο γιο μου ε, ψωνίζει από το AliExpress. Του αρέσει τουλάχιστον. Ε, τι να πω, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι υπηρεσίες θα προσφέρουν γνήσια προϊόντα και νομίζω πως καμία κυβέρνηση, ούτε μόνη της ούτε όλες οι κυβερνήσεις ε, μαζί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο τους το πρόβλημα. Χρειάζεται να έρθουν στο τραπέζι και οι επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποι αυτοί έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς το πρόβλημα. Και στην τελευταία μας συνάντηση μας ζήτησαν αρκετές χώρες να αρχίσουμε να ε, δημιουργούμε κάποιες καταφυντήριες γραμμές έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν από λίγες μέρες διάβασα ένα άρθρο από τον Γενικό Διευθυντή του Alibaba, ο οποίος έλεγε ότι θα ήταν ε, υπέροχο να υπήρχε μόνο μία ε, πλατφόρμα ε, συναλλαγών στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην γίνει αυτό πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Ήταν σημαντική η συνεισφορά σας και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πεπισμένος ότι ε, αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει για πάρα πάρα πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα ελπίζω. Αυτό φυσικά ε, είναι και το τέλος της δικής μας συνεδρίασης, επόμενη συνεδρίαση 11 και 12 Ιουλίου.